πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Περίοδος 2014-2015. Τον λόγο έχει η συγγύρια, συγγύρια πρώτη πρώτη και έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά κυρία μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συγγητές με τους οποίους είχαμε ένα σωρό επικοδομικές συζητήσεις και συνεδριάσεις, αλλά και όλους τους πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν κάποιες προτάσεις που έδωσαν για το ψήφισμα και έχουμε ε, επίσης την υποψήφιση του σχεδίου κειμένου στο site του κόμματος μας του Τσίνκο Στέλλε. Είναι ένα αξιόλογο το κείμενο του ψήφισμα και είμαι ικανοποιημένη γιατί έτσι θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια και έτσι θα εμπλακούν περισσότερο οι πολίτες ε, στο έργο των θεσμικών οργάνων. Πρόκειται για βήματα προς τα εμπρός. Έχονται διαφτάσει μια ιστορική συγκυρία γιατί τώρα ε, τρεμοσβήνει η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα ε, θεσμικά όργανα. Έχουμε κάποιες αποφάσεις του δικαστήριου πολύ σημαντικές αλλά θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ σημαντική διαφάνεια. Όμως οι λόγοι δεν γίνονται έργα. Πολλές από τις ε, συστάσεις σε διάφορα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου τους κατά το παρελθόν δεν ε, είχαν συνέχεια, δεν υλοποιήθηκαν και αυτό αφορά και την συμμετοχή δημοκρατία και τη διαφάνεια που είναι βασικά θεμέλια της δημοκρατίας και τα αναγνωρίζει η Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, ε, μια που έχουμε θεμέλιο την συμμετοχή δημοκρατία, αυτό είναι το πνεύμα του κειμένου. Θέλουμε επομένως να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό μητρό, στο οποίο να έχουν πρόσβαση για τις αποφάσεις, ε, να έχουν πρόσβαση οι πολίτες, να βλέπουν τον τρόπο ε, και τα αποτελέσματα και τον τρόπο που διατίθεται και να μπορέσουμε να ε, υπάρχει πρόσβαση στην ενημέρωση με ένα κοινό σημείο πρόσβασης μέσω των διαδικτυακών θυρών της Ένωσης και επίσης να μπορούν αυτό να το κάνουν και οι ανάπηροι. Θα πρέπει να υπάρχει επομένως διαφάνεια αλλά γι' αυτό χρειάζεται και προστασία των καταγγελών των υπαλλήλων που θα πρέπει να καλυφθούν με κάθε τρόπο και οικονομικά. Και έχουμε κάποιες ε, σχετικές προτάσεις στα πλαίσια της Δημοκρατικής Λειτουργίας της Ένωσης και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με όλη την νομοθετική λειτουργία, το τι θα γίνει επίσης με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαλόγου που δεν ξέρει τίποτα ο κόσμος αυτό πρέπει να καλύψει και το μητρό των ε, λομπιστών γιατί και από εκεί έχουμε διαρροή κάποιων οργάνων. Θα αναγνωρίζουμε το ότι οι άτυποι ε, τριμμένες διάλογοι θα πρέπει να έχουν περισσότερη διαφάνεια και να ελέγχουν έτσι περισσότερο τι γίνεται οι πολίτες. Όσον αφορά τώρα τα λόμπι, υπάρχει μια πρόταση για να υπάρξει ένα ε, μητρό για αυτές τις ομάδες εθνικών συμφερόντων από σε όλα τα θεσμικά όργανα περισσότερη διαφάνεια των ε, διαπραγματεύσεων που καταλήγουν στις διεθνές συμφωνίες. Όσο γίνεται περισσότερα έγγραφα να μπορεί να δει ο κόσμος. Επομένως, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια για τις ε, ε, ε διαδικασίες η παραβάση, τις ε, προς τα κρατη και να είναι γνωστό το τι, τι διαδικασίες γίνονται, ποιοι είναι κάθε φορά οι δικαιούχοι ε, κάποιων νομοθετικών πράξεων για να μην έχουμε απάτες και έτσι θα ανακτήσουμε την χαμένη αξιοπιστία. Αν αυτά δεν τα προσέξουμε θα ήταν μεγάλο λάθος ε, ε, και θα ωφεληθούν οι εθνικιστές να άρουμε επίσης σύγκρουση και, είχε πει ο, ο Καζαλέτζο ότι θα πρέπει να προσέχουμε ε, την εμπιστοσύνη των πολιτών και τον έλεγχο που θα πρέπει να έχουν. Αλλιώς δεν έχουμε ούτε άμεση δημοκρατία και ω ευρωβουλευτές πιστεύουμε στην ελευθερία για τη δημοκρατία. Θα πρέπει όλοι μαζί να συσπηρωθούμε ούτως ώστε να έχει πρόσβαση ο κόσμος στις πληροφορίες. Ή πρόεδρος. Ε, μιλήσατε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα στο τέλος της παρέμβασής σας. Θα έχετε τη δυνατότητα και με την ολοκλήρωση της συζήτησης να λάβετε για άλλα δύο λεπτά για να παρουσιάσετε τα συμπεράσματά σας και τώρα παρακαλώ την Επίτροπο Γιώργο να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, σύντομοι κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή μας, όπως δεσμεύτηκε ενώπιον του σώματος ο Πρόεδρος Γιούνκερ, έχει καταστήσει την ε, διαφάνεια και την αλλαγή προς τη διαφάνεια πρώτο καθήκον. Είναι καθήκον μας αυτό προς τα εκατομμύρια των πολιτών. Είναι δουλειά μας να κάνουμε είναι καθήκον μας να κάνουμε τη δουλειά μας δυνατόν πιο δημοκρατικά και διαφάνεια. Η Επιτροπή ήδη εφαρμόζει ύψιστα στις προδιαγραφές διαφάνειας, αλλά βεβαίως ε, είμαστε δεκτικοί σε κάθε βελτίωση όπου είναι αυτή απαραίτητη και σκόπιμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το γεγονό ότι το ψήφισμα απευθύνει έκκληση στα μέλη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να ακολουθούν την πρακτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ την δημοσιοποίηση των συναντήσεων των κύριων πολιτικών ηγετών και η Επιτροπή με 10.000 τέτοιων ε, δημοσιεύσεων ε, δίνει στη δημοσιότητα τις ε, συνεδριάσεις που την αφορούν. Αυτό όσον αφορά βέβαια και τις διμερείς επαφές με εκπροσώπους των ε, ομάδων πιέσεως, αρμοδίους για λήψη αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο και επιφερειακούς άρχοντες επίσης έχει μεγάλη σημασία. Ε, περιμένουμε, ε, θα, θα καταθέσουμε λοιπόν μια πρόταση διοργανικής συμφωνίας για υποχρεωτικό μητρό διαφάνεια που θα καλύπτει τα τρία κύρια θεσμικά όργανα και με το στοχο αυτό να αυτόν έχουμε ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση από 1η Μαΐου του 2016 με στόχο την υποβολή προτάσεων στο δεύτερο ήμιση του έτους. Η Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι τα τρία θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στην νομοπαραγωγική διαδικασία έχουν καθήκον διαφάνειας και αυτές οι υψηλές αρχές διαφάνειας και προδιαγραφές αργαφάνειας πρέπει να εφαρμόζονται. Η διοργανική συμφωνία λοιπόν πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει την νομοπαραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για μια συμφωνία όπου η Επιτροπή μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα δεσμεύθηκε δεσμεύθηκαν να βελτιώσουν τη διαφάνεια στις νομοθετικές διαδικασίες και να ε, εγκαθιδρύσουν πρακτικές ε, διατυπώσεις για τις μελλοντικέ και διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αντίστοιχα λοιπόν ε, προβλέπεται και η δημιουργία ενός Μητρώου Διαφάνειας για τις κατεξουσιοδότησης πράξεις κατά το 2017 που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια για τις πράξεις που επηρεάζουν τη ζωή του πολίτη και την, ε, τις εργασίες των επιχειρήσεων. Οι συνομοθέτες καλούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσουν τις προτάσεις της για την πρόσβαση στα έγγραφα, την επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης σε κάθε θεσμικό όργανο σε έγγραφα. Ε, αυτό ισχύει βέβαια και θα πρέπει να ισχύει και για κάθε οργανισμό και αποκεντρωμένη υπηρεσία ε, μεταξύ άλλων, εξακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίζει τις προσπάθειες των συνομοθετών προκειμένου να εξασφαλίσουν κοινό πεδίο συμφωνίας για τις δύο προτάσεις για τον κανονισμό 1049 του 2001 και σε σχέση με την πρώιμη δημοσίευση εγγράφων, Ευρωπαϊκή, με την απόφαση για δημοσίευση εγγράφων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οθετήσει μια πρόταση δημοσίευσης εγγράφων με το Μητρό Εγγράφων Υποστηρίζουμε δε τα δοκιμαστικά πιλωτικά προγράμματα που εισάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την εξασφάλιση ευχερού πρόσβασης σε μη απόρριτα έγγραφα που έχουν σε θέση του ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εν όλο, η επιτυχία αυτού του εγχειρήματο θα εξαρτηθεί από την ε, ανάπτυξη συστήματος διαχείριση των εγγράφων των ε, συνομοθετών των θεσμικών οργάνων και βέβαια την αποφυγή της επικάλυψης στην αρχαιοθέτηση των εγγράφων αυτών. Επίσης πιστεύουμε ότι οι κανόνες που ισχύουν και η πρακτική που εφαρμόζεται μπορούν να εξισορροπήσουν την διαφάνεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση δε με την πρόταση για θέσπιση θεσμού Επιτρόπου για τη Διαφάνεια, ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαν, σας διαβεβαιώ και μάλιστα λυπάται που δεν μπόρεσε να έρθει προσωπικός σήμερα, έχει αρμοδιότητα και διασφαλίζει τη βελτίωση των διοικητικών πρακτικών ως προς την πρόσβαση σε έγγραφα και μπορώ και εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι η διαφάνεια είναι μέλημα πρώτης τάξεως για την Επιτροπή στο σύνολό τη. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ακούσουμε τώρα τους ε, αγορητές των πολιτικών ομάδων. Πρώτα η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Είναι απολύτως ουσιώδης η πρόσβαση στα έγγραφα για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο έργο μας και για να κλείσουν τα κενά ανάμεσα στους πολίτες και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Υπάρχουν λαϊκιστές που θεωρούν ότι οι Βρυξέλλες και το διακηρύττουν αποφασίζουν για τις ζωές των πολιτών. Εδώ το μήνυμα του Λαϊκού Κόμματος είναι καθαρό. Δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε. Δεσμευόμαστε υπέρ της, του ανοιχτού χαρακτήρα των θεσμικών οργάνων και της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Να, να καταφανεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με δημοκρατικό τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ρόλο πρωτοπόρου. Μένει να γίνουν και άλλα πράγματα όμω, και από το Συμβούλιο ζητώ από την Προεδρία να αναλάβει την πρωτοβουλία για να γίνει μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι πράττουν οι εκπροσωποί τους και πώς δαπανούν τα χρήματά τους. Και μάλιστα με τρόπο εύχριστο. Για παράδειγμα, ένας ενιαίος ιστότοπος, όπως ε, η Ευρωπύλη, να μπορεί δηλαδή να είναι στη διάθεση του κοινού για να αναζητεί πληροφορίες οι άνθρωποι να μπορούν να συμμετέχουν και να επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φτάνουμε σε άμεση δημοκρατία. Στην Ευρώπη έχουμε θεσπίσει αντιπροσωπευτική δημοκρατία και βεβαίως ο ανοιχτός χαρακτήρας συμβαδίζει με την ευθύνη. Δεν μιλούμε για Wikileaks ούτε για καταγγέλλοντες του είδους whistleblowers. Ασφαλώς η προσωπική σφαίρα οφείλει να προστατεύεται. Και βεβαίως, Λάουρα, οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει να είναι πιο διαφανείς και οι διαπραγματεύσεις, αλλά χρειάζονται όμως και χώρο και χρόνο για να μπορούν να σκέφτονται και για να παραγάγουν αποτελέσματα. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι να είμαι ανοιχτή στο έργο μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και συνεργασία στην Ευρώπη, διότι αντιμετωπίζουμε κοινέ προκλήσει οι οποίε απαιτούν κοινέ ευρωπαϊκέ απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Τώρα, η κυρία Άννα Χέντ, εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα που το προστατεύουν μάλιστα οι ιδρυτικές συνθήκες. Η έκθεση που συζητούμε αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική ζωή. Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Πρόκειται άλλωστε για τον κανονισμό που ρυθμίζει τα της πρόσβασης στα έγγραφα. Αυτός όμως παρεμποδίζεται ακόμα στο Συμβούλιο. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να επιμένουμε διαρκώς ώστε όλα τα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν απολύτως τον κανονισμό αυτό καθώς και τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει σε αυτόν μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας. Μία καλή πρόταση είναι η θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν τον ανοιχτό χαρακτήρα και την διαφάνεια. Αυτά πρέπει να γίνουν απαραίτητος. Η πρόσβαση στα έγγραφα θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια στα μάτια των πολιτών και σε μια βελτιωμένη διαχείριση τα των, Ευρω... τα των... Ε, συγγνώμη, των της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι σημαντικά αυτά. Σε ό,τι αφορά την διαφάνεια, μπορούν βεβαίως να τεθούν διάφορες ερωτήσεις. Χρειάζεται όμως ενίσχυση και του κοινωνικού διαλόγου για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε εμείς την πρόταση αυτή ώστε να μπορούν να επιλαμβάνουν των θεμάτων αυτών με πρόσβαση στα έγγραφα οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Για παράδειγμα, οτιδήποτε έχει σχέση με τον κοινωνικό διάλογο, πρωτόκολλα, πρακτικά δηλαδή και ούτω καθεξής. Αυτά όλα πρέπει να είναι ανοιχτά. Εμείς θα ταχθούμε σαφώς υπέρ της εκθέσεως, δίνοντας έτσι ένα καθαρό μήνυμα ότι κάνουμε κάθε το δυνατόν για να ενισχύσουμε την διαφάνεια στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική ζωή. Η κυρία Μακοβέη. Η Dreptul Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δικαίωμα πρόσβαση στα ε, έγγραφα αλλά και στι πληροφορίε είναι θεμελιώδε δικαίωμα σε οποιαδήποτε δημοκρατία. Διότι απόντω αυτού του δικαιώματο δεν υπάρχει δημοκρατία αλλά δικτατορία. Ο κόσμο έχει δικαίωμα να ενημερώνεται και χρειάζεται να ενημερώνεται σε σχέση με το πώς ε, δαπανώνται τα χρήματά τους, τι γίνεται όσον αφορά την διοίκηση, τι γίνεται την ε, νομοθεσία και όλα αυτά ισχύουν για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να ξέρουν επίση τι πολιτικέ εμεί αποφασίζουμε στο όνομά του. Αυτό σημαίνει νομιμότητα για μα, αλλά σημαίνει και ε, υπευθυνότητα για μας στα πλαίσια του δημοκρατικού συστήματος. Χρειάζεται διαφάνεια επομένως πρόσβαση στις πληροφορίες και έτσι έρεται αυτό το κενό εμπιστοσύνη που υπάρχει τώρα μεταξύ των ε, Ευρωπαίων και των θεσμικών οργάνων. Γιατί πάρα πολλοί πολίτε δυσπιστούν προ τα θεσμικά όργανα, οπότε α του δώσουμε τι πληροφορίε και α άρουμε αυτό το κενό εμπιστοσύνη. Κάποιοι συνάδελφοι ερώτησαν γιατί θα πρέπει ε, στο website να έχουμε όλε αυτέ τι πληροφορίε που δεν χρειάζεται ο κόσμο. Η απάντηση είναι α το κάνουμε και ο κόσμος α διαλέξει ποιε πληροφορίες χρειάζονται και ποιες δεν χρειάζονται. Αυτοί να και όχι εμείς. Για την άλλη, η κυρία είναι τη Ευχαριστώ πρόεδρε και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τα κατάφερε καλά. Ήμουν ε, εισηγήτρια για την προηγουμένη έκθεση που φτιάξαμε πάνω σε αυτά. Μιλούμε για εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη τώρα είναι ε, όσο χειρότερη, όσο, όσο λίγη γίνεται. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε και εμείς τους πολίτες και φαίνεται σαν να μην τους εμπιστευόμαστε γιατί κάνουμε σαν να φοβόμαστε το τι κάνουμε και παρά όλα αυτά τα ωραία που λένε τα τρία θεσμικά όργανα ακόμα δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα το ανοιχτό και της διαφάνειας υπάρχει τάση κρυψίνιας, ε, θέλουμε να δείξουμε όσο γίνεται λιγότερα και ξέρω ότι σας λέω ότι έχουμε να περάσουμε από τα χίλια κύματα για να φτάσουμε σε κάποιες ε, ε πληροφορίες. Έχω πάει δύο φορές στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Επίσης, ε, ο κανόνας είναι η διαφάνεια. Και αυτό δεν είναι κουβέντες φιλελεύθερου. Αυτό είναι ό,τι προβλέπεται από το δίκαιο. Δεν είναι να διαλέγουμε τι θα αποκαλύψουν, να λέμε ότι δεν πρέπει, ας το σκεφτούμε. Η διαφάνεια είναι μια νόμιμη υποχρέωση. Αν δεν θέλουμε διαφάνεια, θα πρέπει κανείς το απόρριτο να το δικαιολογεί. Και ε, αναφερθήκαμε και στο ψήφισμα ε, το οποίο είχα την τιμή να συντάξουμε από δύο έτη. Δεν έλαβε και μια σοβαρή συνέχεια εκείνη μου η και όταν δεν μιλούμε για τη διαφάνεια στους τριμερείς διαλόγους, τότε θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά που κάναμε το 2014. Άρα χρειάζεται να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια τώρα παρά τότε. Τώρα το 16 παρά τότε το 14 γιατί τώρα υπάρχει το κενό εμπιστοσύνη. Επίση τι πρέπει να κάνουμε που τα λέγει και το προηγούμενο ψήφισμα. Να υπάρχει σε όλα τα δεσμικά όργανα κάποιο ε, υπάλληλο για την διαφάνεια. Το έχουμε πει για το Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος πάντα λέει όχι. Επίση ένα πρόγραμμα δράσης κλείνω Πρόεδρε και κατά τρίτο λόγο χρειαζόμαστε κάποιου κανόνες για την διαβάθμιση των εγγράφων και λιγότερη γραφειοκρατία όσον αφορά την αμφισβήτηση της διαβάθμισης για να μην να πάμε δικαστήριο. Σα ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Η κυρία Λιόλ Γκουφμαν ένα παράδειγμα και έτσι μπορούμε να δούμε πόση διαφάνεια υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ κρατώ αυτή την δήλωση που υπογράψουμε για να μπούμε ε, σε κάποια αίθουσα όπου υπήρχαν τα έγγραφα για το TTIP και μας είπαν ότι θα πρέπει αυτό να γίνει γιατί ήταν εκεί διαβαθμισμένα έγγραφα. Επομένω, έτσι είπανε, υπάρχει ασφάλεια για τα έγγραφα και με τίποτα, δεν με πράξη ή παράληψη, δεν είναι δυνατόν κάποιο που δεν έχει ε, άδεια να μην μάθει. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε τα έγγραφα και τις πληροφορίες τους. Και όταν εμείς υπογράψαμε αυτήν την δήλωση, μας είπαν ότι εάν αυτοί οι δεν τηρηθούν θα υπάρξει πειθαρχική δίωξη ή και δίωξη ενώπιον των δικαστηρίων. Δηλαδή μας δείξανε τα έγγραφα με τον όρκο της σιωπής. Μιλάμε για μια επίθεση χωρίς προηγούμενο ε, γιατί τώρα μιλούμε για τις δημοτεύσει με τις ίπα, γιατί τώρα οι πολυεθνικές υπαγορεύουν αυτή τη συμφωνία TTIP όμως απαιτούν ε, τη σιωπή εμείς απαιτούμε δημοψήφισμα για να μιλήσει ο λαός ε, Greens Group ε, Senor Paria κ. Χωσέπ Τερικάμπρας για τους Πρασίνους. Πράσινη, πράσινη αλήθεια. Ε, σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή η έκθεση, ούτω ώστε να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο. Μιλάμε για τη διαφάνεια που θα πρέπει να είναι θέμα προτεραιότητα στην Ευρώπη. Και οι πράσινοι θεωρούμε ότι το πιο σωστό θα ήταν να υπάρχει ένα επίτροπο αρμόδιο για τη διαφάνεια και για την πρόσβαση του κόσμου στα έγγραφα. Έχω τρία στοιχεία να αναδείξω σε αυτήν την έκθεση. Πρώτα πρώτα, το μοναδικό σημείο πρόσβαση από τις διαδικτυακέ πύλες Ευρωπαϊκή Ένωση Δεύτερον, πόσο σημαντικό είναι να δημοσιοποιούνται όσο γίνεται περισσότερα έγγραφα μέσω του ίντερνετ. Επίσης και τα έγγραφα των διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες για θέματα εμπορικά ή οποιασδήποτε άλλη φύσεως. Τρίτον, το υποχρεωτικό μητρό για τα λόμπι. Και εκεί θα κατονομάζονται αυτά τα λόμπι που ασκούν επίδραση στη διαμόρφωση του κοινωτικού δικαίου. Και λέμε στην έκθεση ότι θα πρέπει η Επιτροπή να ε, να ε, έχει μια γενική πολιτική για την διαφάνεια και ευχαριστούμε την συγκέντρια για το έργο της. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Ε, εμείς ευχαριστούμε για το έργο. Ευχαριστούμε για όλα όσα είπατε, ο για των Πρασίνων και τώρα για το EFTT. μισή θα κυρίως Μπάτερν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, Πάντα μιλάει για διαφάνεια, για δημοσιότητα, για έλεγχο από τους πολίτες που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί. Ένα ζήτημα που απασχολεί όλο τον κόσμο είναι η TTIP, η προτινόμενη συμφωνία εμπορικών σχέσεων και επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Την TTIP την διαπραγματεύονται εν και κλειστό, και παραβίστο, δεν έχουν ούτε οι ευρωβουλευτέ τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τι διαπραγματεύσει ή να ελέγξουν την έκβαση αυτών. Μέχρι και 20.000 email έχω λάβει μέχρι σήμερα από πολίτε ψηφοφόρου που ανησυχούν για τη TTIP, η οποία θα επηρεάσει τι δημόσιε υπηρεσίε, την Εθνική Υπηρεσία Υγεία ε, και θα τις αφήσει έρμεα στις μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις. Χρειάζεται ένας μηχανισμός ο οποίος θα επιτρέπει ε, προβλέπει μάλλον ένα μηχανισμό ο οποίο θα επιτρέψει σε διεκτικά δικαστήρια να στρέφονται οι επενδυτέ και ει βάρο ακόμη κυβερνήσεων, εάν αρνούνται αυτέ να ε, ταχθούν στις απαιτήσεις τους. Ε, ο πρόεδρος Ομπάμα την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα απίφθινε απειλές κατά των Βρετανών εάν τυχόν και φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το δημοψήφισμα που πρόκειται να διεξαχθεί τον Ιούνιο. Πόσο χαμηλά μπορεί να έχει πέσει, μας έρχεται εμετός η Βρετανία για να τολμάει κάποιος να της δίνει μαθήματα τέτοιου τύπου και ο Πρωθυπουργός της να μην αντιδρά. Έτσι λοιπόν, ανα πάσα στιγμή θα πρέπει να αποχωρήσουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι θα πρέπει να περιμένουν ε, οι Αμερικανοί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μείζον εμπορικό εταίρο ε, των ΗΠΑ χωρί εμπορική σύμβαση. Παρα, παραγνώρισε ο πρόεδρος Ομπάμα το γεγονό ότι ένα από του μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου ε, το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρω... Ευρωπαϊκή ενώ δεν έχει ειδική εμπορική συμφωνία και όταν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε σχέση με τις εμπορικές μας ε, συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Ο Ομπάμα θέλει να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θέλει να επιβληθεί το TTIP σε όλους μας οι Εβραίοι. Πρέπει να σταματήσουν να αυταπατώνται. Δεν έχουμε ιδιαίτερη προνομιούχο σχέση με τους Αμερικανούς, μόνο δουλική σχέση με τις ΗΠΑ. Το Αμερικανικό establishment δεν είναι φίλοι του, ε, της Βρετανίας του ενδιαφέρουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και τα συμφέροντα του διεθνούς κεφαλαίου. Προς ε, το συμφέρον λοιπόν του Βρετανού πολίτη είναι στις 23 Ιουνίου να, καταψη... υπερψηφίσει την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσει την εφαρμογή της απόφασης αυτής το χειρότερο δυνατό. Ευχαριστώ Ρίτσαρτ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. η κυρία Κατρίνα Κνίτσι. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τη συνάδελφο Φεράρα για τη δουλειά τη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η υπόθεση αυτή για τη διαφάνεια των θερμικών οργάνων πέραν των όσων προβλέπουν οι συνθήκες ε, αυτά δυσκολεύονται για την πρόσβαση οι πολίτε όσον αφορά τα έγγραφα για την νομοπαρασκευαστή λειτουργία και να καταλάβουν επίση τη διοικητική λειτουργία. Και αυτό παρά το ότι δεν υπάρχει κάποιο είδου συντονισμένη προσέγγιση. Το σχέδιο ψηφίσματος τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια για την δραστηριότητα των θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ε, πρότυπο ενίας ε, Αντιμετώπιση και ρυθμίση και άρα έχει σωστή κατεύθυνση. Τώρα περνάμε μια ρίση και νομίζω ότι το να υπάρχει εγγύηση γνώση και ελέγχου της δραστηριότητα των θεσμικών οργάνων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να βοηθήσει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου και να έχουμε εγγύηση της δημοκρατικής συμμετοχής, οπότε γι' αυτό θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να κρατηθούν προς αυτήν την ρότα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, συνάδελφε Ρούχονεν Λέρνεν, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ την κυρία Φεράρα για την πολύ καλή δουλειά της. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική όταν έχουμε να κάνουμε κοινέ αποφάσεις. Δεν αρκεί όμω μόνο η διαφάνεια. Πρέπει να είναι ευχερής η πρόσβαση στις δημόσιες αυτές πληροφορίες. πληροφορίε αν ένας δημοσιογράφος εκπροσωπός με κυβερνητική οργάνωση θέλει να βρει έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να αποφεληθεί από αυτά και να τα αξιοποιήσει εάν ε, αυτά είναι προσβάσιμα δύσκολα από περίπλοκες διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν και αυτή η ευχαίρης πρόσβαση να ληφθεί υπόψη ε, στην έκθεση Φιφεράρα. Άλλωστε αυτό έχει εξασφαλιστεί γιατί μιλάει για καλύτερη πρόσβαση στα έγγραφα. Υπάρχουν βεβαίως όρια στη διαφάνεια. Κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών όπως ε, της TTIP δεν είναι δυνατόν να σε όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή γιατί αυτό θα ε, θέτει σε μειονεκτική θέση τη διαπραγματευτική ε, ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εξασφαλίσετε μια, ένας ελάχιστος βαθμός διαφάνειας απαραίτητος και για την εμπιστοσύνη του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο μας λείπει. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Λόπες Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ε, ε, από ό,τι φαίνεται, ο λόγος που το συζητούμε αυτό το ζήτημα είναι η έκθεση για την πρόοδο στα ε, έγγραφα κατά την περίοδο 14-15 και νομίζω ότι πάρα πολύ καλά τα πήγε η, η συντάκτη και οι σκιώδες. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για την ομορφιαστική διαδικασία, για τους θεμέλιους διαλόγους, γιατί θα πρέπει όλα να είναι εδώ πέρα διαφάνεια, αλλά επίσης θα πρέπει να γίνεται και μετάδοση από το ίντερνετ όσον αφορά τους διαλόγους για την ε, νομοπαρασκευαστική λειτουργία, γιατί θα ε, πρέπει να διαμαρτυρηθούμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει αυτό ε, το οποίο λέμε στην Ισπανία ότι πες μου τι, τι λες και θα καταλάβω τι σκέφτεσαι Οπότε γιατί στην πρακτική δεν ισχύει η χάρτα των δικαιωμάτων. Είναι απαραίτητο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να απεμπλοκεί η χρήση του γενικού δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα. Αυτό μπλοκαρίστηκε στην προηγούμενη θητεία και αυτό θα πρέπει να επιληθεί τώρα. Μα μη κινήσεις ένα λεπτό, Πρόεδρε. Κύριε Γιώργο, αγαπητοί συνάδελφοι. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκληρώσης και της ε, εγκαθίδρυσης των θεσμών στηριζόταν πάντα στην ιδέα της συμμετοχικής δημοκρατίας και της διαφάνειας. Είναι λοιπόν ε, μη πρέπον θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου και του Κοινοβουλίου, να διατηρούν απόρριτα έγγραφα ακόμα να μην εξασφαλίσουν την πρόσβαση αυτά. Το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο και όλα τα νέα σώματα και υπηρεσίες που συζητήσαμε ακολουθούν τον ίδιο κανονισμό της ίδιας για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις και τις διαπραγματεύσεις σε διεθνείς συμφωνίες ισχύει το ίδιο. Είναι πολύ απλό λοιπόν πρέπει εκείνοι οι οποίοι ε, διαθέτουν ως φορολογούμενοι την χρηματοδότηση για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό πρέπει να γνωρίζουν εάν και κατά ποιο τρόπο επηρεάζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία η ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριοι συνάδελφοι, κύριε συνάδελφε. Και τώρα περνάμε στη δικασία Καριστία. Ο κύριος Καπούτο. Presidente. Generare Η γενική προστιθέμενη αξία των εγγράφων από τα κράτη-μέλη για τα ευρωπαϊκά όργανα είναι κάτι το οποίο έχει πολιτικό βάρος, αλλά είναι και κάτι το οποίο άπτεται της εφαρμογής των δημοκρατικών διαδικασιών. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει μια καλύτερη γνώση αυτών των διοικητικών διαδικασιών μέσω της ανοιχτής πρόσβασης σε αυτά κάθε δικαιοδοσία και κάθε ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από την άλλη πρέπει να προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα σε σχέση με τον σεβασμό της ιδιωτικότητας, σε σχέση με την πρόσβαση στα έγγραφα και την ταξινόμηση, τον διαβάθμιση καλύτερα των εγγράφων. Στην πραγματικότητα ε, η όρια αυτή είναι κάτι το οποίο αλλάζει συνεχώς λόγω ακριβώς της χρήσης της ψηφιοποίησης και είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο κώδικα. Είναι λοιπόν απαραίτητο για τις διαδικασίες τριγωνικού διαλόγου για τις ε, τροπολογίες της Ολομέλειας να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες αντιπροσωπευτικοί της δημοκρατίας. Τώρα esis vuleftis, notis Marias, enas lepto παρακαλώ. Ξανά στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε για διαφάνεια, πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, όταν εμείς ως ευρωβουλευτέ μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα της διαπραγμάτευσης ttip υπό τον όρο υπογραφής εγγράφων εμπιστευτικότητας σε ένα δωμάτιο που δεν επιτρέπεται να κρατούμε σημειώσεις ή να φωτοτυπούμε τα έγγραφα όταν δεν μα επιτρέπεται να δημοσιοποιήσουμε το περιεχόμενο των εγγράφων τη ttip. και όλα αυτά όταν οι γερουσιαστές στις ηνωμένες πολιτείες δεν έχουν αυτούς τους περιορισμούς όταν οι βοηθοί τους έχουν και αυτή πρόσβαση στα έγγραφα της ttip όταν επιπλέον 700 εμπειρογνώμονες που δουλεύουν για τη γερουσία τον ηπα έχουν επίσης πρόσβαση στα έγγραφα της ttip μια συμφωνία που ο πρόεδρος ομπάμα ζητά να ψηφιστεί αρωνάρων. μια σύμβαση η διαπραγμάτευση της οποίας είναι η αποθέωση της μυστικής διπλωματίας. για ποια διαφάνεια μιλάτε κυρία Γιουρόβα για ποια δημοκρατία μιλάει η ευρωπαϊκή ένωση όταν οι τρόικες και τα μνημόνια παραβιάζουν τα εθνικά συντάγματα τις ευρωπαϊκές συνθήκες και ανατρέπουν δημοψηφίσματα αδιαφορώντας για τη λαϊκή κυριαρχία. το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στο το μοναδικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες έχει χρέος να πρωτοστατήσει στο δημοκρατικό αγώνα για διαφάνεια και έλεγχο των θεσμών. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, ε, ε, Αντώνιο Μαρίνιο Επίντο. Σας ευχαριστώ, ο Πίντο, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ε, συγχαίροντας ε, την εισηγήτρια, την κυρία Φεράρα. Η διαφάνεια έχει μεγάλη σημασία για τα συμφέροντα των πολιτών μας ε, που όλοι θέμε εδώ πέρα να προστατεύσουμε. Βεβαίως διαφάνεια σημαίνει ευκολία πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες για να προστατευτεί η συμμετοχική δημοκρατία. Τα θέματα λοιπόν και τα προβλήματα πολιτικής ε, διαφάνειας ε, είναι οι εχθροί της ε, δημοκρατίας ε, και των θεσμικών οργάνων. Η πρόσβαση στα έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του εσωτερικού τριμερούς διαλόγου. Στη χώρα μου θα λέγαμε ότι αν δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. Σας ευχαριστώ, Ιβαν Γιάκοβτσιτς. <laughs> Mm, ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ και για την ευγένειά σας απέναντι σε όλους εμάς εδώ. Θέλω και εγώ να υποστηρίξω την εισηγήτρια. Ο στόχος της τελικά είναι οι πολίτες να νιώσουν πιο κοντά στα θεσμικά όργανα και να μπορέσουμε να εργαστούμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ε, να μπορούν να μας ελέγχουν οι πολίτες. Αυτό λοιπόν είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχουν οι πολίτες και μέσω της άσκησης του δικαιώματος αυτού θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους προς τα θεσμικά όργανα. Δυστυχώς τα προβλήματα υπάρχουν, η γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ ισχυρή και φοβάμαι ότι η λέξη διαφάνεια δεν είναι πάρα πολύ σωστή. Αυτό το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το να προσπαθήσουμε να είμαστε δεκτικοί, ανοιχτοί και να τους δίνουμε τις πληροφορίες που επιθυμούν. Ο κύριος Χρυσόγονος. Η πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους τα ευρωπαϊκά όργανα είναι θεμελιώδους σημασίας η εμπιστευτικότητα των εγγράφων θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. αυτό συνάγεται τόσο από τις διατάξεις του σχετικού κανονισμού όσο και από την περιοριστική ερμηνεία που έχει δώσει το δικαστήριο της ένωσης στις εξαιρέσεις που προβλέπονται σε αυτόν. εν τούτης παρατηρούμε πολύ συχνά το φαινόμενο τα ευρωπαϊκά όργανα να αρνούνται στους πολίτες την πρόσβαση σε έγγραφά τους καταστρατηγώντας την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης. χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διατλαντική συμφωνία ttip καθώς ελάχιστες πληροφορίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας λόγω του απόρριτου χαρακτήρα των σχετικών εγγράφων. οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να στραφούν άμεσα προς μια κοινή πολιτική ανοιχτής πρόσβασης στα έγγραφα ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχική δημοκρατία η διαφάνεια και η λογοδοσία απέναντι στους πολίτες. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ε, Κατρίνα Κόνετσνα. Η κυρία Κόνετσνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, έκθεση αυτή. Καταλαβαίνω βεβαίως πως έπρεπε να είστε κάπως διπλωματικοί ε, και ήσασταν βεβαίως ε, ήπια. Ίσως πολύ ήπια. Εγώ δεν θα έλεγα πως ε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο στην διαφάνεια. Μάλιστα η έκθεση της DM25 απευθύνεται στο Συμβούλιο και την Κομισιόν ότι οι Ευρωβουλευτές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα. Παραδείγματο χάρη τα έγγραφα της TTIP δεν μπορούμε να τα δούμε. Και κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε και ε, έγγραφα για την Εξεταστική Επιτροπή. Ελπίζω λοιπόν να συνεργαστούν εδώ πέρα θεσμικά όργανα, αλλά ανήσυχο. Λοιπόν, υπάρχει και το θέμα του κεντρικού μητρώου για τους λομπίστες, το οποίο θα πρέπει να ισχύει όμως για όλα τα θεσμικά όργανα, γιατί ήταν στο τίτι περισσότεροι λομπίστες από ΜΚΟ. Μάλιστα, ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αρχή της διαφάνειας που θα πρέπει να ισχύει στην πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των κοινωτικών θεσμικών οργάνων είναι από τις αρχές που απλώς να καλοποιήσουν ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα συστηματικό αποκρυφισμό και στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου όπως τη ΣΥΤΑ, το ΤΙΖΑ, το ΤΙΤΙΠ χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξοικείωσης με το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Ε, σκάνδαλα ε, όπως το LuxLeaks ε, με τα έγγραφα που συναντήθηκαν επίσης δεν ήταν προσιτά, ούτε καν στους ευρωβουλευτές. Οπότε φαίνεται ότι αυτές οι αρχές υπερισχύουν του δημοκρατικού ελέγχου και της κανονικής διαφάνειας που θα πρέπει να υπάρχει ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, σε θέματα ακόμη και τραπεζικής υποπτίας. Ακόμη και οι ευρωβουλευτές δεν έχουν ε, πρόσβαση σε τέτοια έγγραφα, όπως φάνηκε αυτή τη βδομάδα στην Πορτογαλία. Οπότε ουσιαστικά η διαφάνεια είναι ένα αδιαφανές γυαλί σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επίτροπος η κυρία Βέρα Γιώροβα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και την υποστήριξη που επιφυλάξετε στην αρχή της διαφάνειας. Κάτι που αισθενιζόμαστε απόλυτα. Μάλιστα, στις 2 Μαΐου έχουμε μια εκδήλωση υπέρ της διαφάνειας που θα συμβάλλει στις δημόσιες διαβουλεύσεις για τη θέσπιση του Μητρώου Διαφάνειας που θα καταγράφονται οι ενδιαφερόμενοι στις Βρυξέλλες και ε, πέραν τη Ευρωπαϊκή. Ένωση. Ό,τι αφορά την, ε, τον, την μεταρρύθμιση του κανονισμού, ε, αυτό ακρεμεί στι διαπραγματεύσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να βρουν κάποιο κοινό, κάποιο κοινό έδαφο συνεννόηση. Εν ώψη αυτού του αιτήματο, ε, οποιαδήποτε αίτηση για πρόσβαση ε, συνάδει με τα άρθρα 41 και 42 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τηρήσει και την ομολογία του Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων σε ό,τι αφορά τα έγγραφα που αφορούν έρευνε επί παραβάση που έχουν ε, ξεκινήσει εις βάρος των κρατών μελών. Και προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων και Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διαφορμόσουμε το μέλλον του Μητρώου διαφάνεια. Θεωρούμε ότι σε θέματα όπου υπάρχουν κοινοτικέ αρμοδιότητες για τη διοίκηση, υπάρχει ένα ε, ευρύ πλέσμα, πλέγμα συγγνώμη, κανόνων, αρχών και πρακτικών. Θα πρέπει βέβαια να πιστούμε αν υπάρχει ανάγκη για ειδική ε, νομοθεσία που θα προσφέρει ένα ε, οριζόντιο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου σε αυτό το στάδιο. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα η συγκεκριά μας, η κυρία Λάουρα Φεράρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και κυρίως να ευχαριστήσω τους Κιώδης. Η διαφάνεια είναι ο τελικός στόχος τον οποίο θα πρέπει να πετύχουμε, είναι ένα μέσο για να καλύψουμε την απόσταση ανάμεσα στους πολίτες και τα ευρωπαϊκά όργανα, για να εμπλέξουμε περισσότερο τους πολίτες στην λειτουργία της συμμετοχικής δημοκρατίας. Υπάρχει κοινή γνώμη η οποία φαίνεται να διστάζει σήμερα απέναντι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και άκουσαμε δυστυχώς με λύπη ότι πολλοί πολίτες ε, δεν κατανοούν τα έγγραφα και πολύ συχνά δεν ενδιαφέρονται και να κατανοήσουν τα έγγραφα αυτά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες εγγράφων που δεν προκαλούν κάποιο ενδιαφέρον Και σε αυτό μπορεί να οφείλεται επίσης και στον τεχνικό χαρακτήρα και στην ορολογία η οποία είναι πολλές φορές ε, κατανόητη. Συνεπώς λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτείται να είναι πιο αναγνώσιμη η λειτουργία τους και έτσι <clears throat> θα μπορέσουν οι πολίτες οι ίδιοι να καταλάβουν πού βρίσκεται το συμφέρον τους και πού ανταποκρίνεται η προσοχή τους. Απαιτείται λοιπόν να υπάρχουν πληροφορίες περισσότερες, πληρέστερες και γι' αυτό απευθύνω την έκκληση να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό τόπο πρόσβασης για να γίνει ακόμα περισσότερο σεβαστό το δικαίωμα στην ενημέρωση. Θα πρέπει επίσης να γίνεται ενημέρωση και για την επιρροή των λόμπις, όπως επίσης και για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που γίνονται πολύ συχνά ε, μέσα σε πλήρες σκότος. Συνεπώς λοιπόν η έκθεση αυτή όπως και τα προηγούμενα χρόνια έχει σαν στόχο την διαφάνεια. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση.